Ještě eh, Κυρίε και κύριοι, να ολοκληρώσουμε την ε, συνεδρίαση τώρα και επισήμως τη ε, Υποεπιτροπής ε, Ασφαλεία και Αμήνη, διότι στην συνέχεια, σύμφωνα με τη διάταξη, έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ένα είναι το σημείο που θα συζητηθεί, ένα το θέμα που θα συζητηθεί και αφορά κάποια έκθεση ιδιαίτερη πρωτοβουλίας για τις συνταγματικές νομικές και δεσμικές επιπτώσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε επομένως αυτήν την ε, έκθεση, ε, αυτή η έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού πρόκειται να συνταχθεί από κοινού από τις δύο επιτροπές. Οπότε γι' αυτό και θα κάνουμε κοινέ ε, συναντήσεις και θα είναι κοινό το χρονοδιάγραμμα και θα γίνει μία μόνη και μόνη κοινή ψήφιση της, του κειμένου. Τώρα, οι συνεισηγητές είναι δύο συνάδελφοι. Ο Μίχαελ Γκάλερ από πλευράς Επιτροπής Άμυνας και ο κύριος Γκονσάλε Πόν για την Συνταγματική Επιτροπή. Και οι δύο καλωσορίσατε στην συνάντησή μα. Στη συνέχεια πρόκειται να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή των Προπολογισμών. Και εκεί θα αναλάβει με την γνωμοδότηση αυτή ο κύριος Ζων Αρτουή. Λοιπόν, τώρα να αρχίσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ, οι δύο συνεισηγητές, Γκάλερ και Γκονσάλες Πόνς, να λάβουν το λόγο. Ας μιλήσει πρώτος όποιος θέλει. Διαλέξτε εσείς. Κύριε Γκάλερ. Με ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Γκονσάλες Πόνς, είναι καλό που έχουμε εδώ μια κοινή συνεδρίαση γιατί πρόκειται για μια έκθεση η οποία ε, έχει βαρύτητα και για τις δύο εκθέσεις, ε, και για τις δύο επιτροπές. Το θέμα είναι οι συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνες. Είναι ένα θέμα που δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο. Και βεβαίως κάτω από την εντύπωση των, του αποτελέσματο των Αμερικανών, Αμερικανικών εκλογών. Αυτή τη συζήτηση στη δική μας επιτροπή την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Και θα ήθελα να σας παραθέσω μια φράση του Προέδρου της Επιτροπής ε, ε, χθες. Είπε ο κ. Γιούγκερ θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την άποψη ότι οι Αμερικανοί είναι μέχρι ιστοδυναικές υπεύθυνοι, αρμόδιοι για την, για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ε, και πραγματικά συμφωνώ μαζί του και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό εδώ να εξετάσουμε πως ε, χωρίς να προβούμε σε μια αλλαγή των συνθήκων, κάτι που είναι δύσκολο και σύνθετο, να πώς θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνος. Και νομίζω ότι γενική, το γενικό πνεύμα αυτής της έκθεσης ε, να πούμε ότι ως κινητήρια δύναμη στον τομέα της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι για την ε, συνεργασία με τον συνάδελφο κύριο κονζάλες και επίσης για την συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες εδώ στη ΣΕΝΤΕ, ΑΦΕΤ και ΑΦΚΟ που ε, στηρίζουν αυτό το πρόγραμμα. Ε, το, η έκθεση ε, επικεντρώνεται στα θεσμικά όργανα τα οποία ήδη έχουμε ή θέλουμε να διαμερφώσουμε μελλοντικά όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και ζητήματα προϋπολογισμού στους, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, της κοινή πολιτικής. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια στρατηγικά ζητήματα, όχι τόσο σε ζητήματα ε, λειτουργικά της ε, καθημερινής ε, πολιτικής. Γιατί αυτά τα ακούσαμε από τον κύριο Πάσκου αυτή η έκθεση στηρίζεται, ε, είναι μια έκθεση που ακολουθεί την έκθεση του κυρίου Μπρεσό και Πρόκ ε, που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας, ε, που αφορούσαν την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή επίσης είναι μια έκθεση μετά από τις εκθέσεις της ΕΝΤΕ, όχι μόνο αυτής της θητείας, αλλά και της προηγούμενης που μέχρι στιγμής είχαν πλατιά υποστήριξη από τις πιο διαφορετικές μεταξύ τους πολιτικές ομάδες. Οι περισσότερες από τις ιδέες που έχουν ε, παρουσιαστεί από την είπατε εκπρόσωπο της Επιτροπής και, και από τις χώρες μέλη ε, έχουν εφαρμοστεί και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ορθό και εν ώψη των ε, εξελίξεων αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε σε αυτές, να επανέλθουμε σε αυτά τα αιτήματα και σε αυτές τις βασικές ιδέες και να τα διατυπώσουμε εκ νέου. Όσον αφορά τις ε, συνταγματικές πτυχές ε, αυτής της έκθεσης, θεωρώ ότι υπάρχει ελλειπής δέσμευση εκ μέρους των χωρών μελών για να αξιοποιήσουν την ε, ε, ε, διαρθρωμένη μορφή συνεργασίας. Υπάρχει επίσης μια, μια λυπή σαφήνεια στο Συμβούλιο αλλά και στις χώρες μέλη σε σχέση με το πώς πράγματι θέλουν να ξεκινήσουν αυτή την κοινή πολιτική και να την εξελίξουν περαιτέρω την κοινή ε, άμυνα ε, το άρθρο 42.2 του κανονισμού. Ε, θα πρέπει να διευκρινιστούν θέματα επί παραδείγματι το πώς χρηματοδοτείται η κοινή πολιτική βάσει του άρθρου 41α και πώς μπορεί να διευρυνθεί σε, άλλους, σε άλλα θεσμικά όργανα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα κατά πόσο οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται ε, με ειδική πλειοψηφία βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση από τον ε, Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Προπολογισμό. Ε, ε, στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ε, δυνατότητα εθνικού βέτο. Ωστόσο, ε, ούτως ώστε και οι χώρες που έχουν διαφορετική άποψη να πρέπει να συγχρηματοδοτήσουν. Και ε, ενδεχομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει δυνάμεις σε σύγκρουση με τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία είναι αρμόδια σε εθνικό επίπεδο. Και θα πρέπει να, διευκρινίσουν, να διευκρινίσουμε ότι ποια είναι σύμφωνα με το άρθρο 41α της συνθήκης η χρηματοδότηση των ε, λειτουργικών τμήματων της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Ε, το να μην γίνεται μια τέτοια χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών εν γέννη αυτή είναι μια ε, ανασταλτική, ε, περιορισμένη ερμηνεία, εάν θέλετε, του άρθρου 41α ε, του κανονισμού. Και επειδή τα περιθώρια ερμηνεία είναι ασαφή και επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην νομική υπηρεσία, εμείς ως Κοινοβούλιο ζητήσαμε να υπάρξει μια διαλεύκανση, μια διευκρίνηση μεταξύ των, από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Το άρθρο 179 της Συνθήκης είναι η νομική βάση για την χρηματοδότηση της έρευνας για την άμυνα. Ε, και όχι το άρθρο, το άρθρο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καλύψουμε ε, και είναι το άρθρο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να ε, καλύψουμε με τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλους τους τομείς της έρευνας και όχι μόνο τον τομέα της άμυνας. Υπάρχει και το άρθρο 187 για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά μία συγχρηματοδότηση και εκ μέρου των ε, επιχειρήσεων ε, στον τομέα της ε, άμυνας. Θα πρέπει η Κομισιόν να τα επενεξετάσει όλα αυτά, κάτι που, το, που δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Υπάρχει και το άρθρο 36 της συνθήκης, το οποίο μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί, το οποίο έχει εφαρμοστεί πλήρως ε, και το άρθρο αυτό λέει, θα το αναφέρω στα αγγλικά, ότι εκπληρώνει το έργο της να εξασφαλίσει ότι οι αντιλήψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνονται υπόψη της Επιτροπής. Και πράγματι ε, εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, βελτιώσεις. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ο περιορισμός του θεσμικού ρόλου των, ε, της Επιτροπής Ασφαλείας, της πολιτικής ομάδας, της ομάδας πολιτικής ασφαλείας. Ε, δεν θα έχει κάποιο ρόλο στις, ε, στην εσωτερική ε, δεν θα έχει καθοριστικό ρόλο για την ΚΕΠΑ. ότι εκπρόσωπος μέχρι στιγμή σε σχέση με τη χρηματοδότηση και τον κανονισμό που αποτελεί τη νομική βάση για την υπηρεσία αυτή και αυτό ήταν ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι λένε ότι η συνέχιση της αρχικής νομικής βάσης του 2004 δεν είναι συμβατή με τη συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημεία που κατά την άποψή μου θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση και θεωρώ ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκονθάλεθ. πρώτα πρώτα. τον αγαπητό συνάδελφο Μίκαελ Γκάλερ για την συνεργασία, αλλά για το έργο το οποίο επετέλεσε. Πάρα πολύ σωστά ε, είπε όσα είπε για να συνεισφέρει στην έκθεση. Επίσης ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους της Συνταγματικής Επιτροπής. Ε, και έτσι, επομένως, προωθούμε την έκθεση αυτή. Οι δύο βασικοί άξονες τώρα που αφορούν αυτή την έκθεση είναι η εξή. Δεν είναι δύσκολο να ε, τα ε, αναφέρουμε, αλλά είναι δύσκολο να τα αναλύσουμε. Πρώτα-πρώτα δηλαδή ότι έχουμε περισσότερες δυνατότητες άμυνας. 28 φορές παραπάνω. 28 προϋπολογισμούς άμυνας. 28 νέους διάβλους ε, πληροφοριών. Επομένω, τώρα θα πρέπει και εμεί να πολλαπλασιάσουμε και τι προσπάθειέ μα όσον αφορά την άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είμαστε μακριά από το να εκμεταλλευτούμε όλε αυτέ τι νέε δυνατότητε ε, που προανέφερα για πληροφόρηση, για, για την επιχειρησιακή δυνατότητα κλπ. κλπ. Να τι αξιοποιήσουμε δηλαδή. Άρα επίση, ο δεύτερο άξονα της έκθεσης είναι ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί συντονισμού. Με, με αυτούς μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Όμω δεν αξιοποιούμε τους μηχανισμούς αυτούς. Εάν επομένω τώρα ε, βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει το Συμβούλιο, δεν υπάρχει μια συνολική ε, στρατηγική πολιτική άμυνας για την Ευρώπη, ε, αν θέλουμε επίσης να προωθήσουμε την ε, αρχή της κοινή ασφαλείας, το, πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε τα συστήματα που ήδη ισχύουν, που ήδη έχουμε εγκρίνει, αλλά δεν τα αξιοποιούμε. Οπότε αυτές οι μεταρρυθμίσεις από πλευρά της συνθήκης Λισαβόνας είναι εκείνες που θα πρέπει να είναι καθημερινές γραμμές, ώστε να έχουμε μια τέτοια δομή άμυνας και ασφαλείας. Κοινή Εάν δεν υπάρχει βούληση από πλευρά των κρατών μελών, τόσο ώστε να ενεργοποιήσουμε αυτού του ήδη υπάρχοντε μηχανισμού, ε, τότε δεν έχει νόημα να μιλούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση τη Άμυνα. Ούτε είναι δυνατόν κανένα να ξεκινάει την οικοδόμηση των σπιτιού από τη στέγη. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε με, την, με τη σειρά κάνουμε τα, αυτά τα βασικά και μετά να πάμε πιο μακριά. Επομένω, σε αυτή την έκθεση προσπαθούμε να αναλύσουμε το νομικό πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν προβλεφθεί και δεν χρησιμοποιούνται για την κοινή άμυνα. Και γι' αυτό αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναλύσουμε το άρθρο 42, τη ρήτρα δηλαδή ε, αμοιβαία αρρωγή και βοήθεια και το άρθρο επίση 46 την ενισχυμένη συνεργασία που είναι το άρθρο 20, όλα αυτά είναι παραθέματα από την Συνθήκη της Λισαβόνας και επίσης να δούμε και την συνεργασία ε, που προβλέπει, συνεργασία κάποιων μελών που προβλέπει το άρθρο 44 είναι επομένω προ έκπληξη του ότι τη σήμερα ημέρα με τα, όλα όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, τα, τόσα έχουν γίνει και, και, εκτό, γύρω-γύρω μα. Αυτή η ρήτρα ε, τη ε, αμοιβαία αρρωγή δεν χρησιμοποιείται. Να, είχαμε τι επιθέσει στο Παρίσι. Ε, εντάξει, εκεί την επικαλέστηκαμε, αλλά τα, όλοι οι άλλοι μηχανισμοί δεν έχουν ε, διερευνηθεί. Οπότε θα πρέπει, είπατε, εκπρόσωπος και τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι συνθήκες. Ιδίω όσον αφορά αυτή τη ε, δομή της μόνιμης συνεργασίας, τόσο ώστε να υπάρχει μια κοινή άμυνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος Γκάλερ, κατόπιν των χθεσινών εκλογικών αποτελεσμάτων στη ΣΥΠΑ είδαμε ότι από τώρα η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι λίγο περισσότερο μόνη στον κόσμο. Η Συνταγματική Επιτροπή επίση πρόκειται να αναλύσει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, διότι συνήθως μιλάμε για περισσότερη συνεργασία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αλλά το θέμα της εθνικής κυριαρχίας ήταν ένα βασικό επιχείρημα ή αντεπιχείρημα και ένας φραγμός από τα κράτη ώστε να μην ισχύσουν τα άρθρα της συνθήκης Λισαβόνας που αφορούν την ασφάλεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι με αυτή την έκθεση θα πρέπει να προωθήσουμε τις δύο ιδέες. Πρώτα απ' όλα για μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας ε, δεν είναι κάτι το συμβαστό με την ιδέα της ε, εθνικής κυριαρχίας. Και δεύτερον, να προωθήσουμε το ότι δεν υπάρχει καλύτερη άμυνα της εθνικής κυριαρχίας από το να προστατεύσουμε την εδαφική ακυρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τον ρόλο του Εθνικού, των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος πρωταγωνιστικός. Αλλά δεν θα σταθώ ε, εις αυτό, διότι τα εξήγησε τόσο καλά ο Μάικλ Γκάλερ. Και να κατακλείδη θα πρέπει να σας παραπέμψω σε τρεις πολιτικές ε, συστάσεις που κατά τη γνώμη μου επίσης θα πρέπει να περιέχονται στην έκθεση. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να είμαστε υπέρ του να γίνει κάποιο διάλογο για άμυνα και ασφάλεια ή στο Συμβούλιο. Και να υπάρχει επίση ευρωπαϊκό εξάμεινο μέσου, ούτω ώστε το θέμα αυτό να τύχει η προτεραιότητα σε όλα τα θεματολόγια. Κατά δεύτερο λόγο, επίση, θα πρέπει να είμαστε υπέρ του να έχουμε μια λευκή βίβλο για ασφάλεια και άμυνα. Και πέραν του να προβληματιστούμε για τι στρατιωτικέ ε, δυνατότητε των σημερινών κρατών μελών, να αναλυθεί τι είδου συνεργασία χρειάζεται, τι είδου ε, ε, επιχειρήσει μπορεί να η Ευρωπαϊκή Ένωση τι δυνατότητες μπορεί να υπάρχουν, τι, και, και, και, πόρους, και πόροι, τι χρειάζονται και που θα τους βρούμε. Άρα χρειάζεται να γίνει και μια διοργανική συμφωνία, ούτως ώστε να προκύψει ε, μια πραγματική ουσιαστική συμφωνία, συμβασμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και μια τέτοια κοινή πολιτική αμήνας και ασφάλειας δεν μπορεί να είναι το σύνολο των επιμέρους πολιτικών των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστό χάρτης πορείας που να στηρίζεται στις ισχύουσε συνθήκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Ο κύριος Τροζιεύσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχά σε δύο πράγματα που είπαν οι εισηγητέ μας, ο κύριο Γκάλερ και ο κύριο Γκονζάλε Πόν. Ο κύριο Γκάλερ στην παρέμβασή του μας είπε το ακόλουθο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο υποεξέταση ζήτημα. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο δεν προβλέπει συγκεκριμένη εφαρμογή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Υπάρχει ένα σαφέ έλλειμμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται και τι βέλτιστε πρακτικέ. ανεξάρτητα μετά όσα λέγονται στην υφιστάμενη έκθεση. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ενισχυτικό, να το πω διαφορετικά. Έχουμε ήδη πολύ καλέ εκθέσει γνωμοδοτήσει, έχουμε διεξάγει καταπληκτικέ συνεδριάσει και συνδιασκέψεις. Αλλά όταν μιλάμε για εφαρμογή, τότε α το πούμε ξεκάθαρα, μιλάμε για πραγματική καταστροφή. Στο τέλος τους στο τέλος των παρεμβάσεών τους οι εισηγητές είπαν ότι ε, η πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι το σύνολο των εθνικών πολιτικών άμυνας και ασφάλειας. Μα συμφωνώ με αυτό. Με άλλα λόγια δεν έχουμε μια κοινή ενιαία πολιτική ασφάλειας και άμυνας η οποία θα είναι σε θέση να υπερβαίνει τις εθνικές πολιτικές άμυνας και ασφάλειας. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια νέα πολιτική. Είναι σημαντικό γιατί πολύ φοβάμαι ότι μία ακόμα φορά θα εγκρίνουμε με ευρία πλειοψηφία ένα κείμενο, το οποίο όμως δεν θα οδηγήσει σε συγκεκριμένη εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Με άλλα λόγια και το νέο κείμενο δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη πρόοδο. Επίσης, πολύ φοβάμαι ότι με τις εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον νέο πρόεδρο μπορεί να βρεθούμε κάπως απομονωμένοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι θα συνεργάσετε πλέον τόσο πολύ μαζί μας σαν ω πρόεδρος των ΗΠΑ. Επίκυνται και άλλε εκλογέ, Αυστρία, κάτω χώρε, Γαλλία και πολύ φοβάμαι ότι στις εθνικές αυτές εκλογές δεν θα δούμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα συμβάλλει στο αίσθημα ασφαλείας και σταθερότητας που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια λοιπόν στιγμή πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε ίσως από την αρχή, να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι κάνουμε στη ΣΕΔΕ τι κάνουμε στην ΑΦΚΟ, τι κάνουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να διασφαλίζουμε κάθε φορά ότι όντως σημειώνουμε πρόοδο, ότι όντως ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών. Αναλωνόμαστε σε θεωρητικές συζητήσεις, αλλά δεν προχωρούμε σε έμπρακτη εφαρμογή των όσων αποφασίζουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι συνδιασκέψεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ κατέληξαν σε πολύ ωραία συμπεράσματα και αποτελέσματα. Περνάει όμως ένα χι χρονικό διάστημα, δεν γίνεται τίποτα στην πράξη και επαναλαμβάνουμε στη συνέχεια μέσω εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια απουσία στρατηγική, μια απουσία στρατηγική προσέγγιση, μια απουσία ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Σα υπενθυμίσω λοιπόν για μία φορά ακόμα ότι η εργασία που κάνουμε εδώ, που κάνουν συγκεκριμένα οι συγγητέ μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, να μην αρχιοθετηθεί σε κάποιο συρθάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σντρογεύσκη. Θέλει να πάρει το λόγο κάποιος από τους και συγητές τώρα. Η κυρία Μπρέσο. Ο σκιώδης εισηγητής μας δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα, συμμετέχει στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Θα ήθελα εγώ σύντομα να αναφερθώ στις δικές του παρατηρήσεις και να βασιστώ στα όσα είπε ο συνάδελφος Γκάλερ, ο οποίος είπε ότι θα βασιστεί στην εργασία που κάνω εγώ και ο Μπρόκα και ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς βέβαια αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να μπούμε σε πραγματικές λύσεις των προβλημάτων που έχουν τοπιστεί. Η δική μας έκθεση, αν θέλετε, είναι λίγο πιο θεωρητική. Πρώτη παρατήρηση. Όντως θα πρέπει να ακούσουμε τα όσα μας λένε οι δύο εισηγητές στις παρεμβάσεις τους. Αναμφίβολα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη ευαίσθητη στιγμή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του πλανήτη θα έλεγα. Και μολονότι προφανώς θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια ειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα μπορεί να συνεργάζεται ειρηνικά με τον υπόλοιπο κόσμο, βλέπουμε παράλληλα ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε κι εμείς ένα σύστημα αποτελεσματικής ασφάλειας. Αυτό προβάλλεται ως ανάγκη όλο και περισσότερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλές εκκλήσεις ως προς αυτό, με μηδαμινά όμως αποτελέσματα σε επίπεδο κρατών μελών. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, προκειμένου και τα ίδια τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν πως έχει κατάσταση αναλάβαμε εμείς μια πρωτοβουλία η οποία προέρχεται από τη Γερμανία και από τη Γαλλία, μια πρωτοβουλία στην οποία έχει συμμετάσχει και η Ιταλία, η οποία ακόμα δεν έχει υποβληθεί επίσημα. Ακούσαμε και κάποιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από την ύπατη εκπρόσωπο. Με άλλα λόγια βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει μία κάποια πολιτική διεργασία για να αντιμετωπίσουμε τελικά ένα ζήτημα το οποίο μέχρι στιγμής το είχαμε αφήσει μόνο στο εθνικό επίπεδο, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ιδίω στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και βέβαια οι πρόσφατες αμερικανικές εκλογές επιταχύνουν την πολιτική αυτή ανάγκη παρέμβασης πλέον από εμά στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα είχε πει ότι περίμενε πλέον από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τα μεμονωμένα κράτη της, περίμενε μία μεγαλύτερη συμμετοχή στην ε, κοινή πολιτική άμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί το ΝΑΤΟ με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι είναι απολύτως αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της. Και προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό αν τα κράτη-μέλη πρώτα δεν αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Μέσω, όπως το είπαν και οι συνάδελφοι, όχι μέσω μιας εγκατάλειψης της εθνικής κυριαρχίας τους, αλλά μέσω μιας αύξησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους μέσω της μεταφοράς κάποιων αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να έχει μια πιο ενισχυμένη πολιτική άμυνας και ασφάλειας, το οποίο συνάδει απόλυτα με τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν, ακόμα και τα πιο σημαντικά και τα μεγαλύτερα, να δρούν μεμονωμένα. Και αυτό το βλέπουμε και στις σχέσεις που έχουμε με τη Ρωσία και στις σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία. Δεν μας το υπενθύμισε αυτό δηλαδή μόνο ο Ομπάμα και ο Τράμπα, αλλά και άλλοι διεθνείς παράγοντες ή άλλες χώρες ή άλλοι πρόεδροι όπως η Ρωσία και η Τουρκία σε όλες αυτές τις χώρες, αλλά και στις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, δεν μπορούμε να προβαίνουμε σε μια μεμονωμένη πολιτική. Από τη μια λοιπόν υπάρχουν οι πολιτικές ανάγκες και κλήσει, από την άλλη υπάρχουν και οι ίδιοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες συμφωνούν πλέον ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ευρεία πολιτική άμυνας και ασφάλειας πάνω από το 70% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι ο τομέας της άμυνας και της ασφάλειας είναι ένα σημαντικό επί του οποίου θα πρέπει να αναλάβει ευρύτερη δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι υπάρχει ή επίσης, ίσως επειδή ακριβώ υπάρχει ένας αναδιόμενος σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για αυτόν τον λόγο προβάλλεται ως όλο και πιο επίγουσα ανάγκη να έχουμε μια ευρωπαϊκή πραγματική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Προφανώς θα πρέπει να περάσουμε από διάφορα στάδια. Προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα πρωταρχικό στάδιο ενισχυμένης συνεργασίας και συντονισμού, να καταφέρουμε δηλαδή από κοινού να συντονίσουμε την αμυντική μας έρευνα, θα πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά τα απαραίτητα στάδια που θα μας οδηγήσουν σε μία ενίσχυση των αμυντικών μας ικανοτήτων, σε συλλογικό όμως επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προτάσεις που κάνουν οι δύο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, να έχουμε ένα μοντέλο ευρωπαϊκού εξαμήνου για την άμυνα, πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε καλύτερα και με τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία οφείλουν και αυτά να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούνται για κάτι τόσο σημαντικό που τελικά επηρεάζει τη δική τους εθνική πολιτική άμυνας και ασφάλειας και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική γνήσια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Εμείς και στην έκθεση που συντάσσω μαζί με τον συνάδελφο Μπρόκ έχουμε ήδη εντοπίσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα θεσμικά πλαίσια, υπάρχει θεσμική βάση. Αν αρχίσουμε λοιπόν να επιτελούμε την εργασία αυτή, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πραγματική ολοκλήρωση, η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό. Και εκεί όμως πάλι πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια θεσμικά στάδια. Δεν γίνεται όμως να τα καλύψουμε εν μία νυχτή, προκειμένου να καταφέρουμε να δρεώσουμε πρώτα συντονισμό και να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό, θα πρέπει να δούμε σε ποια άρθρα τη συνθήκη πρέπει να βασιστούμε και ποια προβλήματα ενδεχομένω να προκύψουν. Καθήκον μας πάντως είναι να καταδείξουμε καταρχάς ότι υπάρχουν τα νομικά εργαλεία και ότι μπορούμε πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ πρόσφατα μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός της άμυνας και της ασφάλειας. Επομένως βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί. Το Συμβούλιο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του Συμβουλίου η ειδική πλειοψηφία. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο της χρηματοδότησης και αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί βάσει της εξής αρχής. Όσοι εμπλακούν στο όλο εγχείρημα θα πρέπει και να το χρηματοδοτήσουν. Στη συνέχεια, Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πιο πολύπλοκο ζήτημα της ε, υποχρέωσης χρηματοδότησης, συμβολής μάλλον στη χρηματοδότηση, ακόμα και από τις χώρες εκείνες οι οποίες θα αποφασίσουν τελικά να μην συμμετάσχουν σε αυτή τη διαρθρωμένη αμυντική συνεργασία. Νομίζω πάντως ότι και αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένουμε με μεγάλη υπομονησία την έκθεσή σας. Hvala lijepa. Kolege prije mene su govorile o širim kontekstu, Širim kontekstu. Αγαπητοί συνα... Α, οι συνάδελφοι ε, απευθύνθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ή μάλλον μίλησαν για ένα ευρύτερο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης σε αυτό το γενικότερο επίπεδο μπορώ να πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αν δεν έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήμα ε, δυσκολεύεται πάρα πολύ να ορίσει την ε, εξωτερική της ε, πολιτική. Θα μένω στον τίτλο αυτής της έκθεσης «Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της, κοινή, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας». Μέσω αυτών των πέντε άρθρων του κανονισμού της συνθήκης είναι σαφές ότι έχουμε την ε, βάση για την ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών. Το άρθρο 42 λέει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια προδευτική ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Επίσης ε, αναφέρεται σε μια βαθμία βελτίωση των στρατιωτικών μας ε, δυνάμεων, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Επίσης ορίζονται δυνατές μορφές συνεργασίας, ε, συμμαχίες εκείνων που θέλουν να συμμετάσχουν και η άλλη δυνατότητα βεβαίως είναι η συνεχής διαρθρωμένη συνεργασία. Επίσης έχουμε άλλα άρθρα το 45 ή 46 που αναφέρονται λεπτεριακά με το πώς ε, θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και ποια θα πρέπει να είναι η νομική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Και στην περίπτωση τις συμμαχίες του συνασπισμού δηλαδή και στην περίπτωση της α, ε, μόνιμης διαφρομένης, της συνεχιζόμενης διαφρομένης συνεργασίας. Επίσης ορίζονται τα καθήκοντα ενός ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας και αναφέρεται το ζήτημα της εναρμόνισης των προμηθειών, του συντονισμού της έρευνας κλπ όλοι οι στόχοι οι οποίοι ε, διατυπώθηκαν το 2008 όσον αφορά τις ε, κοινέ προμήθειες και την κοινή έρευνα δεν έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί και εντωμεταξύ από το 2008 Έδαμε με ένα περιορισμό των κοινών δραστηριοτήτων ή της κοινή ε, έρευνας αυτών τον τομέα η συμμετοχή στην EDA δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 27 ε, μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν εδώ. Όλα όσα είπα καθιστούν σαφές ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν θεσμικά ή συνταγματικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ε, όταν συζητούμε αυτή την έκθεση και ίσως θα έπρεπε να φωτίσουμε περισσότερο ποια είναι τα ουσιαστικά προβλήματα και εμπόδια. Γιατί 15 χρόνια μετά την ε, απόφαση να διαμορφωθεί κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Ε, Εμείς σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η κοινή έκθεση ήταν κάτι που αποφασίστηκε πριν το αντυχές Brexit και πριν την εχθεσινή εκλογή του Ντόνατ Τραμπ ως νέο πρόεδρο τον είπα 20 Ιανουαρίου θα λέω τα Οπότε έχουμε αυτά τα δύο τρομερά γεγονότα τα οποία έχουν πάρα πολλές σοβαρέ και δεν μπορούμε να τα δούμε αποστασιοποιημένα σε σχέση με την ε, έκθεση και όπως γνωρίζετε. Ε, εγώ ήθελα να μείνουμε κατά την εκστρατεία για τον Brexit, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε και τώρα θέλω να έχουμε όσο γίνεται πιο soft αποχώρηση. Ε, να προστατευτεί κυρίω η οικονομία μας στο Λονδίνο και τώρα έχω μια μελέτη που συγγράφω επ' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση της άμυνας και της ασφάλειας. Ε, ο Τραμπ είναι κατά του ΝΑΤΟ, κατά της, του, των πολυμερών ε, πολιτικών και επομένως ε, το τι θα κάνουμε σε αυτούς τους τομείς είναι πολύ σημαντικό. Και κατά τις διαπραγματεύσεις ε, για το Brexit θα πρέπει να δούμε πώς θα μείνει κοντά στην Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά. Βέβαια, εμείς είμαστε πυρηνική δύναμη και έχουμε τις πιο αποτελεσματικές όπλες δυνάμεις στην Ευρώπη και εμείς και οι Γάλλοι. Οπότε, δυστυχώς, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση του 48 με τη συνθήκη των υπαραισίων είναι κάτι το οποίο προηγήθηκε τη συνθήκη της Ρώμης που ίδρυσε την ΕΟΚ και αυτό είναι κάτι το οποίο καλύφθηκε τελικά τη συνθήκη της Λισαβόνας τότε ε, θεωρήθηκε ότι ε, καλύπτεται και δεν χρειάζεται τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό μια που θα φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να εξεύρουμε νέους ε, τρόπους και να δούμε το πώς η Βρετανία θα μπορεί ως κράτος να ε, είναι μέσα στην εκτονική ασφάλειας και άμυνας. Γιατί νομίζω ότι η περιουσία της Βρετανίας μπορεί να προσφέρει και στρατιωτικά. Έτσι και αλλιώς πρέπει να διαπραγματευτούμε κάποιο παρεδώσει την συμμετοχή μας στην η αγορά. Οπότε ναι, θα έχουμε κάποιες ε, θα συμμετάσχουν σε κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες χώρες άσχετες όπως Νέα Ζηλανδία και Ουκρανία. Οπότε τα, τα, τα έχω συζητήσει και με κάποιον ε, πολύ σημαντικό υπουργό της κυβέρνησής μας με τις διαπραγματεύσεις να βρούμε κάποιο είδους καθεστώς ε, παρατηρητή στην Επιτροπή Ασφάλειας κάτι ανάλογο με πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ και έχουμε Ρωσία και Ουκρανία που έχουν κάποιους ε, πρόσδευτες οι οποίοι συμμετέχουν σε εργασίες του ΝΑΤΟ. Όταν όμως το ζήτησα αυτό ε, και το είπα στους διπλωμάτες δεν ε, υπήρχε και τόσο ενδυσός με την πρότασή μου. Πάντως ε, ξέρουμε ότι ποια ήταν η αντίδραση της Μόσχας για τις αμερικανικές εκλογές. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση, τόσο ώστε να μείνει κοντά στι εδώ μέσα άμυνας ασφάλεια η Βρετανία. Κυρία Λουέζινγκ, έχετε το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο Τσαρλ. Στάνοκ. Δεν είναι η σειρά μου. Okay. Okay. Ich teile... Ε, Συμμερίζομαι ορισμένες ε, ε, σκέψεις οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα από την εκλογή του Τραμπ. Το θέμα είναι τι είδους συμπεράσματα, τι είδους συμπεράσματα θα πρέπει να φωτίσουμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ένα συμπέρασμα είναι ότι η ακραία, τα ακραία λαϊκιστικά κινήματα ενδυναμώνονται. Και πέρα από τα βασικά θέματα που αφορούν στρατιωτικοποίηση κλπ. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ε, Φέρνουμε ωστόσο μια μεγάλη ευθύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τους όρους με τους οποίους διεξάγουμε εδώ τη συζήτηση και το, τις προτεραιότητες που δίνουμε ένας όρος όπως είναι η εθνική κυριαρχία στην αξιολόγηση όλων αυτών των θεσμικών ζητημάτων περί των οποίων ομιλούμε δεν είναι η ύψιστη αξία. Εγώ ίδια δεν είμαι εθνικίστρια. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι το κοινοβουλευτικό δικαίωμα στην απόφαση, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και ιδιαιτέρως ε, την ε, πολιτική ασφαλείας και άμυνας, ε, σε κανένα άλλο κοινοβούλιο δεν ε, παραγνωρίζοντος εδώ. Είμαι συντονίστρια στη ΣΕΔ εδώ και πολλά χρόνια ε, και δεν θυμάμαι πότε έχουμε έχουμε πει τη γνώμη μας για τέτοια θέματα. Θυμάμαι όταν πρόκειτο να γίνει μια στρατιωτική αποστολή στη Λιβύη ε, τότε κληθήκαμε εμείς ε, οι συντονιστές ε, από τον κύριο Κόλ και το είπαν ότι το Συμβούλιο το αποφάσισε. Αυτό ήταν, αυτό ήταν ο ρόλος μας. κύριε Γκάλερ, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλες πτυχές ενός Ευρωπαϊκού στρατού. Αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με, με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Γιατί εάν έχουμε αυτό το δικαίωμα και αυτό το οποίο κάνουμε δυσετησίως με τις ε, εκδρομές μας στις ε, χώρες ε, της Προεδρίας του Συμβουλίου, αυτό κατά την άποψή μου και όσον αφορά το λεγόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι μια φάρσα. Δεν πρόκειται για κανένα ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γι' αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, ε, παρακαλώ σκεφτείτε το. Θα πρέπει να τορίσουμε συνέχεια το θέμα της εθνικής κυριαρχίας συνεχώς ή θα πρέπει καλύτερα να μιλάμε με όρους κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γιατί εάν οι πολίτες συνειδητοποιήσουν ότι δεν ασκείται απολύτως κανένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, τότε οι ερμηνείες μπορεί να παρεκκλίνουν προς μια κατεύθυνση από την οποία δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επανέλθουμε. Ε, γίνεται λόγος για τη λεγόμενη διαρθρωμένη μορφή συνεργασίας και λοιπά, να ενεργοποιηθεί και λοιπά. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα, πρέπει, δεν θα λαμβάνονται πλέον συνετικές αποφάσεις. Θα πρέπει, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας για τα θέματα εφαρμογής και όσον αφορά τα δεξιά κινήματα σε ορισμένε χώρες, τι θα γίνει στις χώρες αυτές εάν ε, τα κινήματα αυτά ενισχυθούν. Και αυτό αφορά και το άρθρο 43.3. τα θέματα της στρατιωτικής παρέμβασης ότι μπορεί να καθορίζονται μόνο από το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση, μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε πόσο αυτό πόσο πολύ αυξάνουν όλα αυτά την αποξένωση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το βιώνω κι εγώ ίδια. Πόσο δύσκολο είναι ορισμένα πράγματα να τα εξηγήσουμε στους ε, πολίτες, οι οποίοι κατεβάσουν τα νερολά ε, πολύ γρήγορα. Και σκέφτομαι το εξής. Εγώ πραγματικά κάνω σοβαρή προσπάθεια να αυξήσω τη διαφάνεια των διαδικασιών εδώ προς τα έξω και βιώνω το πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσουν στον πολίτη. Αλλά ορισμένα πράγματα ε, δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει. Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς στον πολίτη ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο τελικά. Και όταν πρόκειται για έναν λεγόμενο ευρωπαϊκό στρατό που υπάρχουν πάρα πολλές ε, επιφυλάξεις και ελπίζω ότι ορισμένες από αυτές τις επιφυλάξεις τουλάχιστον να μπορέσουν μέχρι ενός σημείου να συζητηθούν ουσιαστικά από μας εδώ. Ο κύριος Ευχόζερ έχει τώρα το λόγο. Σα ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν σα άκουσα πριν από λίγο. Θα είμαι πολύ σύντομο, διότι δυστυχώ και ζητώ συγγνώμη πρέπει να αποχωρήσω. Εγώ ήμουν σαφώ υπέρ τη Ευρώπη ε, τη άμυνα και μάλιστα κατέβαλα προσπάθειες και όταν συζητούσαμε τη συνθήκη του Μάστρικτ και στην περίοδο που ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της των μεσών της δεκαετίας του 90, το 95, το 2000 εργαζόμουν για την Ντασό, μια μεγάλη αμυντική βιομηχανία της Γαλλίας και συνειδητοποίησα ότι πίσω από την έννοια της κοινή άμυνα δεν υφίστατο κανείς. Κανείς ο οποίος να μιλά για αυτονομία και ανεξάρτητη άμυνα. Μόνο η Γαλλία και η Ρωσία μιλούσαν για το ζήτημα αυτό η Γαλλία η οποία δεν είχε τα απαραίτητα μέσα, θα το δούμε στο, μέσο, και η, στο μέλλον και η Ρωσία η οποία κατάφερε τελικά να γίνει αυτόνομη από πλευρά άμυνα. Για να έχουμε λοιπόν μια κοινή άμυνα θα πρέπει να έχουμε καταρχά ένα κοινό όραμα. Θέλουμε πραγματικά μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπω οι Άγγλοι μα θέλουμε, θέλουμε τελικά μια Ευρώπη η οπω οι αγγλοι μα θελουμε τελικα μια ευρωπη η οποια ειναι υποκειται στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε ουσιαστικά μια άμυνα η οποία έρχεται να συμπληρώσει την άμυνα του ΝΑΤΟ ή θέλουμε να συμπληρώνουμε απλώς τις προσπάθειες που κάνουν οι ΗΠΑ. Εγώ πιστεύω ότι αν μιλάμε για άμυνα θα πρέπει μόνοι μας να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την άμυνα αυτή χωρίς να εξαρτώμαστε από άλλους. Οτιδήποτε διαφορετικό ουσιαστικά υπονο... υπονοεί ότι είμαστε υποταγμένοι σε άλλους οργανισμούς. Όσον αφορά τώρα την ενισχυμένη συνεργασία, αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει από κοινού και δεν το κάναμε τελικά. Να σας υπενθυμίσω την αποτυχία των Eurofighters, ένα πολύ κακό αεροπλάνο, ενώ τα Mirage, τα Ραφάλ είναι σαφώς ανώτερα και στήχησαν και πολύ λιγότερο. Δεν καταφέραμε να έχουμε συγκεκριμένες ανταλλαγές όσον αφορά τα υποβρύχια, διότι είμαστε σε άμεσο ανταγωνισμό με τη Γερμανία στις εξωτερικές αγορές. Δεν καταφέραμε να καταφέρουμε να έχουμε κοινά αεροπλανοφόρα. Είπαμε ότι θα μπορούσε εδώ να συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια κοινή στρατηγική για τα αεροπλανοφόρα. Να αναφερθώ σε δύο τομείς όπου θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Έχουμε ένα Ινστιτούτο Γάλλο-γερμανικής έρευνας στον τομέα της άμυνας στο Σαν Λουί. Θα μπορούσαμε στα πλαίσια του Ινστιτούτου αυτού να καταφέρουμε να συνεργαστούμε προκειμένου να έχουμε αυτή την περίφημη ενισχυμένη συνεργασία που θα ενίσχυε τελικά και το Ινστιτούτο αυτό, στο οποίο εργαζόταν και ο πατέρας μου. Και κάτι ακόμα. Είδα ότι έχει γίνει και μια έκθεση όσον αφορά αυτό το ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος το οποίο απέρριψαν κάποιοι συναδελφοί μου. Μα νομίζω ότι ακριβώς το χώρο αυτό, τον απολογιστικό, τον, στον κυβερνοχώρο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αν δεν μπορούμε εμείς να φτιάχνουμε τα chips, αν δεν μπορούμε εμείς να φτιάχνουμε τα routers, αν δεν μπορούμε εμείς να ελέγχουμε τα δίκτυα, ε, τότε η άμυνα για τον κυβερνοχώρο θα καταρρεύσει. Αν για παράδειγμα έπρεπε να εκτοξευτούν κάποιοι πύραυλοι, μάλλον έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια αεροπλάνα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε την απαραίτητη, τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτή τη στιγμή προκειμένου να προχωρήσουμε σε τέτοιες στρατιωτικές κοινέ επιχειρήσεις. Και οι Γερμανοί μας λένε αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να γίνονται παγκόσμιοι δημόσιοι διαγωνισμοί. Το πρόβλημα όμω είναι ότι θα πρέπει εμείς πέρα από τον εξοπλισμό που έρχεται απ' έξω, να μπορούμε οι ίδιοι να δημιουργούμε τα συστήματα αυτά, να δημιουργούμε αυτούς τους εξοπλισμούς. Γιατί αν μια μέρα, για παράδειγμα, η Γαλλία γινόταν εταίρος μιας ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, αν καταφέρναμε να επιστρέψουμε σε μια Ευρώπη των εθνών, σε μια Ευρώπη ανεξάρτητων εθνών, πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται αν δούμε πώς κινούνται τα πράγματα. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να δούμε πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Αν η, βλέπαμε τις αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας τα τελευταία 30 χρόνια, τότε θα καταλήγαμε όλοι σε πάρα πολύ υψηλό χρέος. Νομίζω ότι έχουμε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρήσεις στην Αφρική, χωρίς όμως να φροντίζουμε τελικά να

θεραπεύουμε του εθνικού μα προπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτόν το λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά που μιλάμε για δημοσιονομική εξυγίανση. Και σαφώ η Γαλλία θα πρέπει να προχωρήσει σε μια δημοσιονομική εξυγίανση. Και σαφώ χρειαζόμαστε και μια χρηματοδότηση. Χίλια δισεκατομμύρια δίνουμε από τη μία μέρα στην άλλη για να σώσουμε τι τράπεζε. Για ποιο λόγο όμω δεν δίνουμε 100-200 δισεκατομμύρια για την κοινή ασφάλεια και προστασία μα στα πλαίσια τη πραγματική οικονομία. Όλε οι επενδύσει στην αμυντική βιομηχανία είναι επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία τελικά και στη μελλοντική μας ικανότητα να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τις θέσεις απασχόλησης. Χωρίς επενδύσεις στην άμυνα δεν θα είχαμε τα ABS, δεν θα είχαμε τα συστήματα αυτόματης έρευνας μέσω ραδιοπλοήγησης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε φορά που επενδύουμε στην άμεση και στην ασφάλεια, ουσιαστικά επενδύουμε στην προηγμένη τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει στη συνέχεια και την συμβατική, αν θέλετε, οικονομία. Κάντε λοιπόν συγκεκριμένε προτάσει. Πείτε ότι χρειαζόμαστε 100 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασία. Ας ξεκινήσουμε όμως από το γαλλογερμανικό αυτό Ινστιτούτο, ας ξεκινήσουμε με συγκεκριμένες έρευνες, για παράδειγμα στον τομέα της προστασίας του κυβερνοχώρου. Αν κάποιος εχθρός μας τελικά ε, εισβάλλει στα συστήματα επικοινωνία μα, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή και με ενημερώνουν οι καλύτεροι εμπειρογνώμονε για το ζήτημα αυτό, τότε τα συστήματά μα είναι άχρηστα, αν δεν μπορούμε δηλαδή να τα προστατεύσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι στη διαχείριση των συστημάτων αυτών και σιγά σιγά σταδιακά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη Άμυνα και ασφάλειας, σεβόμενη όμω την εξαρτησία και την κυριαρχία των κρατών μελών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σαφχόιζερ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Δόντο, έχετε το λόγο. Εδώ, εδώ είμαι. Θα ήθελα από τη συζήτηση να συμφωνήσω. Βέβαια είμαι μέλος της ΑΦΚΟ, δεν είμαι ειδικό, οπότε τι να πω για αυτό που ο κύριος Γάλλος συνάδελφος αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Πρώτα-πρώτα διότι η γαλλογερμανική πρόταση με αφετηρία το Brexit δεν είναι μία σύμπτωση. Νομίζω ότι είναι σαφής αυτή η συγκυρία που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας να μην έχουμε τον μενο Βασίλειο στα θέματα της άμυνας. Αυτό είναι κάτι το οποίο χτύπησε το καμπανάκι του συναγερμού στην Γερμανία. Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι ακολούθησε αυτή εκείνη η πρόταση Μέρκελ Ολάν. Τα είπε και η κυρία Μπρέσο ότι οι Ισπανοί και οι Ιταλοί υπουργοί άμυνας ενδιαφέρθηκαν αμέσω. Και λογικά Στην ίδια πρωτοβουλία πρόκειται να προσχωρήσουν και χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνω τι επιφυλάξει πολλών συναδέλφων τη Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με κάτι το οποίο ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Υπάρχει όμω αυτή η διεθνή συγκυρία που μεταβάλλεται άρδιν. Επομένω, να μια πολιτική ευκαιρία για την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει αυτή την ευκαιρία να τη χάσουμε. Οπότε, και με βάση το τι είναι στη ΣΥΠΑ. Άρα η Ευρωπαϊκή Άμυνα θα πρέπει να αρχίσει να οικοδομείται χωρίς να εξαρτώμεθα από τις ΣΥΠΑ ε, όπως έγινε τα τελευταία 40 χρόνια. Θεωρώ ότι με αυτή την έκθεση αναδύεται η ανάγκη του να συνειδητοποιήσουμε κάτι το οποίο έχει σχέση με τον φετινό προπολογισμό, συνάδελφε, με την γαλλογερμανική πρωτοβουλία και με την επιστολή ε, των Ισπανών και Ιταλών που έστειλαν την Επιτροπή για πρώτη φορά για την επιμόνιση του προπολογισμού δεσμεύσαμε κάποιου πόρου όπως έλεγε ο Γάλλο συνάδελφο και έτσι να υπάρξει έρευνα ε, στα θέματα τη άμυνας ένα πρώτο βήμα έγινε επομένω. Προφανώ βασίστηκαν σε κάποιε στρατηγικέ πληροφορίε. Είναι κάτι επομένω πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιομηχανία. Άρα πρόκειται για μια ευκαιρία η οποία πρόκειται να προχωρήσει τώρα που η Ευρώπη καλείται να αναδιατάξει την εσωτερική ε, θεσμική αρχιτεκτονική οπότε και άμυνα όπως και ασφάλεια είναι τομείς πάρα πολύ σοβαροί πέρα από τις επιμέρους διαφορές μας. Έχουμε διαφορές στην μεταναστευτική πολιτική, στην οικονομική πολιτική, είμαστε πολύ διασπασμένοι, έχουμε το, τη διαφορά, το χάσμα βορρά-νότου, οπότε έχουμε και αυτές τις διαφορές μεταναστευτικού και οικονομικού θέματος. Έχουμε τις διαφορές ε, Δύσης-Ανατολής, Έχουμε τους φεντραλιστές, ε, τους άλλους που είναι λιγότερο φεντραλιστές. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι διαχωρισμοί. Όμως είναι ένα θέμα, ίσως είναι το μόνο, το μόνο που τώρα που ήρθε η ώρα του να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη με, για τις διαπραγματεύσεις του Brexit, ε, το μόνο θέμα που τρόπο θα συζητήσουμε τι Ευρώπη θέλουμε. Μια Ευρώπη που μπορεί και πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια, να προστατευτεί από την τρομοκρατία και την ε, ασφάλεια και με τη γεωπολιτική της διάσταση. Στην ε, ΑΦΚΟ συντάσσουμε και τις εκθέσεις Μπροκ, τις εκθέσεις του κ. Μπροκ για την συνήθεια της Λισαβόνας. Έχουμε επίσης και την έκθεση ε, τα, τα κείμενα του της εκθέσης του κύριου Φερχόφστατ. Όλα αυτά θα έχουν σημασία μετά το Brexit. Άρα να, που κολλάει το θέμα άμυνας ε, ασφάλειας και γι' αυτό και είναι και μια ευκαιρία που παρουσιάζεται. Άρα θα πρέπει να καθισχάσουμε τους ε, σκεπτικιστές. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι πραγματικά μαζί. Και έτσι θα πρέπει να ανατρέξουμε στο πνεύμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρούσαν εκείνοι ότι είναι βασικός πυλώνας ε, του όνειρου που είχαν για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και ασφάλεια. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Κέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ιδίω αν δούμε τι συνέβη με το Brexit και με τις Αμερικανικές εκλογές. Δεν έχουμε λοιπόν καμία απολύτως δικαιολογία πλέον. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας υπάρχει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια θεωρητικά στα εγγραφά και όχι στην πράξη. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε λοιπόν άλλο με την ε, έμπρακτη εφαρμογή της. Θα ήταν ε, εγκληματική αμέλεια να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και χαίρομαι πολύ που οι δύο συνάδελφοι Γκάλερ και Κονζάλε Πόνς μας ε, υπέβαλαν αυτή την πρωτοβουλία υψής της και μας προτείνουν διάφορους τρόπους για να καταφέρουμε τελικά να ελοποιήσουμε αυτή την πολιτική. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τροεύσκη, ότι θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε ένα ακόμα έγγραφο το οποίο θα το αμελήσουμε στη συνέχεια και δεν θα το εφαρμόσουμε ποτέ. Θεωρώ ότι είναι κοινό μας καθήκον η τελευταία αυτή έκθεση που θα συνταχθεί να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε στην πράξη να την εφαρμόσουμε διότι όπως είπαν και οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης, η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει πολλές ευκαιρίες τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να συντονιστούμε πλέον. Πόσοι μηχανισμοί ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Τα πρακτικά ζητήματα της χρηματοδότησης, της έρευνας, της άμυνας, της υποστήριξης της αμυντικής βιομηχανίας πρέπει να επιληθούν. Και συμφωνώ ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας συνάδει με το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα όμως δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς το σύνολο των επιμέρους εθνικών πολιτικών άμυνας. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και συμφωνώ με τον συνάδελφο Κοζάλες Πόνς θα πρέπει να έχει τον δικό της οδικό χάρτη. Και νομίζω ότι ως προς αυτό έχουν ήδη γίνει κάποιες πολύ προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε τον θεσμικό ρόλο της ε, Πολιτικής και Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβλέψουμε πλέον και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα συστηματικό διάλογο για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη που χρειάστηκε να εγκαταλείψω την αίθουσα για λίγο. Ε, Βέβαια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, αυτή η συζήτηση και θα πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τα όσα είπε ο Στάνοκ για την ανάγκη να ε, διατυπώσουμε κάποια συμπεράσματα του Brexit, σε σχέση με το Brexit στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να αναπτύξουμε κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με την συμφωνία που θα αναπτύξουμε με τη Βρετανία γιατί δεν είναι δυνατόν να μην παραμείνει η Βρετανία ε, συνδεδεμένη με μια Ευρώπη ε, ασφάλειας ε, και ακούγεται ηρωνικό γιατί η Βρετανία το ποικοτάριζε αλλά ε, εν ώψη της παρούσας κατάστασης ε, ελπίζω η Βρετανία να συνειδητοποιήσει ότι το χρειάζεται και εμείς το χρειαζόμαστε. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μετά τα όσα είπε η κυρία Λόζινγκ. Το ζητούμενο, το διακύβημα είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Πάντοτε το ουσιαστικό θέμα ήταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, ιδίως όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και εδώ το ζητούμενο είναι ο δημοκρατικός έλεγχος. Και όταν ξεκινήσαμε την υποεποτροπή το 2004, δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι ότι μάθαμε για το για, το, για μία αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κονγκό ε, και το σχετικό αίτημα για την αποστολή αυτή το μάθαμε από τους Γερμανούς συναδέλφους το, από το Bundestag. Έτσι το μάθαμε. Ε, και στη συνέχεια μπορέσαμε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ε, μακρύς ο δρόμος για να φτάσουμε εκεί και καταλαβαίνω αυτό που λέει η κυρία Λέζινγκ. Πώς να εξηγήσουμε ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανένα έλεγχο. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια ε, είναι σε θέση να ασκήσουν ε, ναι, ένα έλεγχο, ίσως το Bundestag, μια εξαίρεση, αλλά το γαλλικό κοινοβούλιο και το δικό μου κοινοβούλιο δεν έχουμε απολύτως καμία δυνατότητα ε, διενέργειας κοινοβουλευτικού ελέγχου, άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ε, γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει αυτή τη ε, δυνατότητα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά τα θέματα αυτά, ώστε να εξασφαλίσουμε να έχουμε μια πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Υπήρξε μια εποχή που το πολιτικό και στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στο ΝΑΤΟ, ε, τελικά μας εμπόδισαν να αναλάβουμε ένα τέτοιο ρόλο και εμπόδισαν κατ' ουσία την Ευρώπη από το να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Ε, ε, το να μην υπάρχουν τέτοιου είδου υπηρεσίε. Θυμάμαι όταν έκανα την έκθεση για την ασφάλεια στην ε, ναυσιπλοεία, που είναι μια σημαντική πτυχή τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, ε, διαπίστωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, για την, ε, για την ασφάλεια στην αυσιπλοεία που η έδρα του είναι στην Λισαβόνα. για την, ακριβώς την εξασφαλή στην ασφάλεια στην αυσιπλοεία είχε εξαιρετικέ αρμοδιότητες. Είχε και τον αντίστοιχο εξοπλισμό και ήταν, θα μπορούσε να παράσχει πολύ ουσιαστικές πληροφορίες για την Ατλάντα. Στην, για την Ατλάντα στην, και τη σχετική αποστολή στην Σομαλία. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιου είδους συνεργασία και αυτό είναι εντελώς γελίο. Οι προσπάθειες που έγιναν να σωθεί τον Γαλιλαίο να εξασφαλιστεί κοινή χρηματοδότηση για τον Γαλιλαίο. Ε, το Γαλιλαίο ε, έχει ευρωπαϊκή διάσταση και δεν είναι δυνατόν ε, να διαχωριστεί από την ε, πολιτική ασφάλειας και την... Πρόκειται λοιπόν για ζητήματα αυτοτέλειας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο της ε, βιομηχανίας, της τεχνολογικής ε, βάσης, της έρευνας, τα όσα είπε ο Μάικλ, ε, το ζήτημα της έρευνας το οποίο συνδέεται με την βιομηχανία. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υποστηρίζονται αυτές οι προσπάθειες και όσον αφορά τον προπολογισμό αλλά και ο, νομίζ, έλεγχος αφορά τον έλεγχο, νομισματικός έλεγχος αφορά τον έλεγχο των δαπανών, γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό διαφθοράς στις στρατιωτικές προμήθειες σε όλες τις χώρες μέλη. Και καμία, κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν ασκεί έλεγχο όσον αφορά τη διαφθορά στις ε, προμήθειες, ούτε καν το Bundestag αλλά θα ήθελα να απαιτήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διενεργήσει αυτό τον έλεγχο ε, κατά πόσο τα κονδύλια ε, χρησιμοποιούνται ε, με ακέραιο τρόπο και πάνε στη σωστή κατεύθυνση στην αγορά του αμυντικού εξοπλισμού και επίσης όσον αφορά τις ε, δυνατότητες διαστρέβλωσης της αγοράς. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικός ο έλεγχος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κοινή Ευρώπη ασφάλειας και άμυνας. Γιατί η εθνική κυριαρχία είναι σημαντική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε από κοινού να κάνουμε ε, αυτό που θεωρούμε αναγκαίο στο επίπεδο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μόνο η κοινή προσπάθεια μπορεί να μας εξασφαλίσει, όχι η εθνική κυριαρχία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κοινή πολιτική σε όλους αυτούς τους τομείς. Και επίσης συμφωνώ με το είπαν ε, οι συνάδελφοι για την κυβερνοασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί μεμονωμένα να εξασφαλίσει αυτή την ασφάλεια. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει και δεν έχουμε τους πόρους. Ε, πάρα πολλά κονδύλια ε, ε, ξοδεύονται άσκοπα, διασπαθίζονται. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική βούληση. Δεν αφορά μόνο την συνταγματική βάση Υπάρχει η πολιτική, ε, είναι και το θέμα της πολιτικής βούλησης, όλο αυτό το χάος στη Λιβύα. Ε, γι' αυτό είμαστε εμείς ε, ευθύνη, γιατί είχαμε σπαταλήσει τις δυνάμεις μας, τις μεταξύ μας διενέξεις, αντί να μεριμνήσουμε για την κοινή μας εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και τις απειλές που ε, προέρχονται από τη Λιβύη, για να μην πω τη Συρία. Τι λύση βρέθηκε για τη Συρία. Οι χώρες ε, ε, ούτε καν προβαίνουν σε αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών ε, για το πού πάνε τα όπλα που ορισμένα από αυτά πάνε στους πεσμεργά, άλλα πάνε αλλού. Ούτε καν ε, τα στοιχεία αυτά δεν ανταλλάσσουμε, δεν το κάνουμε ούτε καν για τη δική μας ε, ασφάλεια. Και εδώ θα έπρεπε πραγματικά να ξεδιαλύνουμε όλο αυτό το πολιτικό χάος. Μια σημαντική, ένα σημαντικό συμπέρασμα, το, το, σημαντικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έδρα της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχουμε ένα 20 το λέει ο Πρόεδρος, αφού ευχαριστεί την κυρία Γκόμες. Τώρα, πριν ξαναδώσουμε στους συνεισηγητές τον λόγο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να πω τα εξής. Να σας παραθέσω από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 42 παραγραφός 2. Η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας θα οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα. Άπαξ και αυτό αποφασιστεί ο ομοφόνος από το Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν κάποια απόφαση σύμφωνα με τόσο προβέντος του Εθνικό Σύνταγμα. Το Δεκέμβριο, σας υπενθυμίζω, θα συνεργάσει το Συμβούλιο. Οπότε θα ήταν καλή ιδέα να λάβουν υπόψη τη δεκαετία του 90 που είχαμε την κρίση στο Κωσυφοπέδιο στα Βαλκάνια και η Ευρώπη δεν μπόρεσε να παρέμβει. Και αντί ημών επιχείρησαν οι Αμερικανοί με την αεροπορία τους. Ίσως αυτό να μην χρειαστεί να γίνει στο μέλλον. Είναι η δική μας μοίρα και η δική μας Ευρώπη και πρέπει να την προστατεύσουμε. Τώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Κονσάλες Πόνς και μετά στον κύριο Γκάλερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο ούτως ώστε να συμβάλλουν. Η ευχαριστώ και την κυρία Μπρέσο. Η δική μας έκθεση είναι συνέχιση από πλευρά αύκο τη έκθεση τη δική τη και του κυρίου Μπρόκ. Ναι, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή η έκθεση και όλοι πιστεύουμε για τον ρόλο αυτής της έκθεσης όμως είπαμε ότι είναι και μία έκθεση που έρχεται τη σωστή στιγμή. Όλοι συμφωνούμε σε σχέση με το ότι κατόπιν των χθεσινών αμερικανικών εκλογών η Ευρώπη είναι πιο μόνη. Οπότε, όπως είπα μονοχάρογη, όχι μόνο χρειάζεται αυτή η έκθεση, αλλά είναι και ε, μια έκθεση που έρχεται τη σωστή στιγμή. Βέβαια τώρα υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Ο στόχος της έκθεσης είναι να δούμε το πόσο αυτό το χάσμα θα γίνει μικρότερο. Ε, εντάξει, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε 100% στα κράτη-μέλη αυτό το οποίο θέλουμε. Αλλά αυτό το που μπορούμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε μια προσέγγιση αλλά πρέπει να έχουμε μια στάση ρεαλιστική. Θα πρέπει πρώτα πρώτα να, διερευνήσουμε τι δυνατότητες παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν έχει νόημα να μιλούμε για κοινή άμυνα, εάν πρώτα πρώτα δεν έχουμε διερευνήσει το τι δυνατότητες ε, προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν αυτές οι λίγες δυνατότητες που προσφέρονται δεν τις εκμεταλλευτούμε, και τότε δεν έχει νόημα να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα. Και γι' αυτό, βέβαια, πρόκειται για κάποια έκθεση η οποία δίνει εντύπωση ότι είναι ακόμα μια έκθεση. Σωστό είναι αυτό. Όμω είπαμε ότι είναι η έκθεση αυτή μια έκθεση που έρχεται τη σωστή στιγμή και που θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση που πρέπει χωρί να, να, να, υπάρχει εναλλακτική, γιατί δεν υπάρχει πρέπει να προχωρήσουμε και ακριβώς συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος Γκάλερ, ότι δηλαδή θα πρέπει τα κοινοβούλια να είναι στο επίκεντρο αυτής της ε, προβληματικής και επίσης πρέπει να είναι το επίκεντρο της ε, κοινή πολιτικής αμήνης στο μέλλον. Και επίσης, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν να εμπλακούν γιατί μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε το να υπάρξει τέτοιο σχεδιασμό στην άμυνα ούτω ώστε να εμπλακούν τα κοινοβούλια. Ε, άρα χρειαζόμαστε σε αυτήν την προσπάθεια και τα εθνικά κοινοβούλια. Επίση συμφωνώ ότι η πολιτική άμυνα είναι αδελφική τη. Ε, άλλη μια πλευρά τέλο πάντων της, ε, Μόνο αν υπάρχει η μία έχει νόημα η άλλη. Ε, ωραία, μπορούμε να κάνουμε όμως μια έκθεση και να μιλούμε για κάποια κοινή εξωτερική πολιτική. Εάν το αποτέλεσμα των Αμερικανικών χθεσινών εκλογών είναι κάτι το οποίο μας κατέριξε ότι χρειαζόμαστε κοινή άμυνα, ε, επίσης το κατέριξε και για το ότι χρειάζεται μια κοινή εξωτερική πολιτική και να μιλάει με ενιαία φωνή η Ευρώπη. Γιατί σε έναν, όλα αυτά γίνονται σε έναν κόσμο που πια δεν θα συμμετέχει, θα έχει αποσυρθεί η Αμερική. Οπότε το πρόβλημα τώρα δεν είναι το πώς θα αναδιατάξουμε τις συνθήκες ή τα θεσμικά όργανα. Το πρόβλημα είναι το να υπάρξει βούληση πολιτική. Τα κράτη-μέλη δεν θέλησαν, δεν θέλουν και ούτε θα θελήσουν κοινή πολιτική ασφαλείας. Εμείς όμως θα πρέπει να τα υποχρεώσουμε να κατευθυνθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση, σε μια πολιτική Ασφάλεια κοινή. Δεν υπάρχει αναλεκτική λύση, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Ε, αυτό λέμε στην έκθεση, ότι χρειάζεται πολιτική βούληση και η οποία πολιτική βούληση όχι απλώ εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Οπότε και συμφωνώ 100% μετά στο είπε κύριο Τάνοκ. Χθε ένα συνάδελφό σα, κύριε Τάνοκ από το δικό σα κόμμα, μου έλεγε ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι νήσος. Δεν είναι σκάφος, δεν είναι καράβι. Και μετά το Brexit δεν πρόκειται να ξανοιχτεί στους ωκεανούς. Θα συνεχίσει να έχει τη θέση της, θα συνεχίσει να είναι γείτονά μα. Επομένω, όλοι εμεί οι οποίοι είμαστε υπέρ του να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει επίση να είμαστε υπέρ του πιο soft Brexit που μπορεί να υπάρξει. Να μην καταργηθούν όλα, να μην φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, μιλώντα για κοινή η πολιτική ασφάλειας ε, δεν θα είναι μια αυθεντική πολιτική ασφάλειας εάν δεν συμμετέχει η Βρετανία για χάρη της ίδιας και για χάρη των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Και κλείνω τώρα πρόεδρε με ε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ραμόν Χάραγη, με τα οποία και συμφωνώ. Και καταλαβαίνω από αυτά τα οποία πολύ καλά εξήγησε το ότι το κάθε κράτος ε, μέλλον δεν μπορεί να... Ε, θα συνεχίσει μάλλον να υπάρχει, γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει ενιαία αγορά. Μπορεί να είμαστε σε χειρότερη θέση, αλλά θα συνεχίσουμε να, να υπάρχουμε. Βεβαίω και χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία. Αλλά και χωρί δημοκρατία θα επιζήσουμε. Όμω, πάρα πολλά κράτη-μέλη είναι σίγουρο ότι στο μέλλον δεν πρόκειται να επιβιώσουν εάν δεν υπάρχει πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Δεν μιλώ για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά πολλά κράτη-μέλη θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν θα μπορούν να επιβιώσουν ε, αν δεν υπάρχει μια τέτοια κοινή πολιτική άμυνα. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε και δίνω το λόγο στον κύριο Γκάλε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με, τα όλα, με όλα όσα είπε ο συνάδελφο κ. Γκονζάλη. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα επαναλάβω. Και φαντάζομαι ότι η έχει δημιουργηθεί ήδη μια συνέδεση για μια λειτουργικά αναπτυσσόμενη ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας θα δημιουργήσουμε μια κοινότητα γιατί δεν έχουμε προχωρήσει σε άλλους τομείς τόσο πολύ ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ε, μια κοινή πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς έχει αναπτυχθεί σε πολλές ε, χώρες μέλη η αντίληψη ότι ας το κάνουμε, ας αναπτύξουμε μια κοινή στάση στην εξωτερική πολιτική και στην, ε, στην, πολιτική, ασφα... στην πολιτική ασφάλειας και στην πολιτική άμυνας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή η συζήτηση για έναν ευρωπαϊκό στρατό. Δεν ε, σχετίζεται με αυτή τη συνθήκη και μας ε, αποσπά την προσοχή από αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε. Είναι σημαντικό το να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ έχω την άποψη ότι μπορούμε να το κάνουμε εάν εξηγήσουμε ε, ποιες, είναι, ποιες μπορούν να είναι οι λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας ε, ή να κάνουμε προμήθειες μέσω της EDA, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, γιατί αυτή είναι που συντονίζει τα προγράμματα και έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε τις διαδικασίες προμηθειών στις οποίες αναφέρθηκε η Άννα. Ε, Εάν ε, λοιπόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο επειδή είναι πιο αποτελεσματική από τις εθνικές υπηρεσίες ενδεχομένως και αν εδώ ε, κινηθούμε από κοινού ίσως μπορούμε να αναλάβουμε και κάποιες άλλες αρμοδιότητες, να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες μας. Ε, τώρα, όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει ε, ε, να, εδώ θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το οποίο κάνει η διακοινοβουλευτική διάσκεψη. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Και νομίζω πρέπει να ενισχύσουμε και την ε, διακοινοβουλευτική συνδιάσκεψη. Ε, όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει προσδεδεμένη σε αυτή την πολιτική. Ε, ένας ε, επικοδομητικά εργαζόμενος παρατηρητής είναι ίσως πιο πολύτιμος από ένα παρακολύοντα από ένα παρακολύον μάλλον μέλος. Ίσως ε, η Βρετανία ως ουσιαστικός ε, παρατηρητής καλή την πίστη να διανοίξει κάποιες διαφορετικές προοπτικές. Το να παρακολείς ορισμένες φορές είναι χειρότερο. Τώρα, όσον αφορά την ε, έρευνα για την άμυνα, να μην γίνει υπάρξουν παρανοήσεις παρακαλώ, αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει σε αυτό το τομέα είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις εθνικές προσπάθειες. Δεν είναι δυνατόν να το κάνει γιατί είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Αλλά το ζητούμενο είναι με την έρευνα για την άμυνα να συνοδεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει για τις διάφορες αποστολές ε, της ε, κοινής πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας. Το ζητούμενο δεν είναι να κοινοτικοποιήσουμε συνολικά την έρευνα για την άμυνα. Εδώ αυτό θα ήταν υπερβολικά μεγαλόπνο, δεν το εννοούσα έτσι. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές. Να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις τεχνικής φύσης. Στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Ε, η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών, η καταληκτική, θα είναι στις 15 Δεκεμβρίου. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσοι συμμετείχατε στην ε, προετοιμασία της σημερινής συνεδρίασης, δηλαδή το προσωπικό, τη γραμματεία, τους βουλευτές, τους βοηθούς τους, ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς, ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό η συνεδρίασή μας, η κοινή αυτή συνεδρίαση των δύο επιτροπών, ΑΦΚΟ και ΣΕΝΤΕ. Η επόμενη συνεδρίασή μας, η επόμενη συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ, θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου, σε 9 η ώρα το πρωί.